Παρασκευή το πρωί ένα λεωφορείο συγκρούστηκε με τοπικά έξω από τον Μπορντό με μία ανταλίκα και τα δύο οχήματα ε, έπιασαν φωτιά και ήταν ένα από τα πιο βαριά ε, δυστυχήματα με λεωφορεία στην Ευρώπη. 43 άτομα έχασαν τη ζωή τους, κυρίω, κυρίως ηλικιωμένοι, οι οποίοι είχαν ξεκινήσει εκδρομή στα Πρινέα και ήταν λίγο έξω από την γενετηρά τους. Και ακριβώς επειδή είμαστε στη Γαλλία εδώ, θα ήθελα εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ευχηθώ γοργή ανάρρωση σε όσους τραυματίστηκαν στο δυστύχημα αυτό και θα ήθελα στους συγγενείς ε, των θυμάτων να εκφράσω τα βαθιά συλληπιτήριά μας. Ευχόμαστε κάθε δύναμη στους συγγενείς τους στις φρικτές αυτές απώλειες που υπέστησαν. Κυρίες και